πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέχρι τότε. Ε, χαιρετίζω την προσοχή ε, και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται και τη σημασία που αποδίδεται στην άμυνα και ε, την ασφάλεια. Τα σημεία 10 και 11 αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό για την έρευνα και την ανάπτυξη και το έγγραφό μας είναι απλώς μία τοποθέτηση, μία γνωμοδότηση, διότι η Επιτροπή Ήτρε ουσιαστικά ηγείται του θέματος. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι τα στοιχεία της ε, άμυνας και της ασφαλείας. Ε, το 10 και 11 είναι τεχνικά θέματα και ουσιαστικά ο εισηγητής δεν έχει προτείνει τροπολογίες στο 810 υπήρχε κάτι αλλά για το 811 δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Η βασικότερη τροπολογία είναι η πρώτη στο 809 που είναι η πλέον σημαντική καθότι λέγεται ότι η έρευνα και η ανάπτυξη στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 δεν θα πρέπει να αναφερθεί μόνο στην πολιτική τεχνολογία αλλά στην διητή ε, εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της ανάπτυξης. Άρα βλέπουμε ότι ε, η άμυνα για μας δεν είναι ένα θέμα οικονομικό. Είναι, ε, υπάρχει μια παγκόσμια αγορά 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 25-30% καλύπτεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή μια μεγάλη, ένα μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο που επηρεάζει την ε, ε, οικονομική ανάπτυξη σε πολιτικό επίπεδο και εκεί ακόμη μπορούμε να επιδείξουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων ε, από διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ευχαριστώ ε, για τα σχόλια του συναδέλφου Μαυρονικόλα. Το άλλο βασικό θέμα είναι η κατάρτιση ενός χωριστού κεφαλαίου για την ασφάλεια και την άμυνα και η Επιτροπή μας θα ήθελε να θέσει το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Εχθές το βράδυ ε, κατέθεσα και εγώ τις δικές μου τροπολογίες. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι εξαιρετική. Έχει πάρα από... Ε, και ε, πιστεύω ότι προκαλεί και πολλές θετικές τροπολογίες. Αντιλαμβάνομαι ότι ο εισηγητής ε, έχει διατυπώσει απολυτικές ε, τροπολογίες και σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω που πρέπει να προσθεθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθώς είστε και εισηγητής θα είμαι ευθύς. Πιστεύω ότι η έκθεσή σας δεν είναι καλή. Πιστεύω ότι βαίνει προς την λάθος κατεύθυνση. Σπάνια λέω κάτι τέτοιο τόσο άμεσα, αλλά πιστεύω ότι εδώ είναι η κατάλληλη περίσταση, διότι αυτό που προτείνεται να κάνουμε είναι να αντιστρέψουμε μια πολιτική που αυτό το κοινοβούλιο έχει διατηρήσει εδώ και πολλά χρόνια. Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται στην έρευνα για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Έχουμε συμφωνήσει στο παρελθόν ότι τα ζητήματα πολιτικής ασφάλειας θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι του χαρτοφυλακίου έρευνας που χρηματοδοτούμε. Και εμένω σε αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Λούχαν ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μια σημαντική αγορά πολλά υποσχόμενη. Δεν έχω αντίρρηση προς αυτή τη διάσταση, ή το να συνεχίσουμε αυτή τη διάσταση στην έρευνα. Αλλά αυτά που προτείνει ο εισηγητής και προφανώς αυτά που προτείνουν και ορισμένοι συνάδελφοι από εδώ τα δεξιά και που θα το υποστηρίξουν ίσως είναι να διευρύνουμε αυτό το πεδίο εφαρμογής και ρητά να ενσωματώσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία την αμυντική έρευνα ως αυτό σκοπό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για λόγους δημοκρατικούς. Πιστεύω ότι δεν υπήρξε ποτέ ευρεία ανοιχτή δημόσια συζήτηση όπου ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την ανάπτυξη θα χρησιμοποιηθεί για την έρευνα και την προμήθεια στρατιωτικών υποδομών. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση για να γίνει μια τέτοια ε, μεταλλαγή. Δεύτερον από οικονομική άποψη. Φυσικά η αμυντική βιομηχανία αναζητά νέους, ε, νέες πηγές χρηματοδότησης, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ πιεσμένη διότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί υπερικόπτονται. Εγώ πιστεύω και γενικά αυτό το κοινοβούλιο πίστευε ανέκαθεν ότι η σωστή απάντηση σε μια τέτοια απέτηση θα ήταν να προωθήσουμε την ατζέντα του pooling and ε, sharing, της κοινή χρήσης, της συγκέντρωσης και κοινή χρήσης, ώστε να αποφύγουμε τις παλιές υπερβολικές δαπάνες και να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη ενοποίηση με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές δαπάνες που έχουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη να γίνουν πιο αποδοτικές μέσω της συνένωσης και κοινής χρήσης του pooling and sharing. Υπενθυμίζω σε όλους ότι στο τέλος της άσκησης ε, όταν, όταν συναντήθηκαν οι υπουργοί Άμυνας ε, είχαν 300 προτάσεις ε, συνένωσης και κοινής χρήσης και στο τέλος ουσιαστικά προσδιορίσαν 12 προγράμματα με τα οποία θα συνέχιζαν. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι υπερβολικά φιλόδοξο και γνωρίζω ότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις εδώ. Ξέρω ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, εκφράζεται περισσότερη πίεση. Η δική μου κυβέρνηση μάλλον προσπαθεί να φρενάρει τα πράγματα παρά να σε αυτές τις προσπάθειες. Αλλά αν αυτή τη στιγμή ανοίξουμε τον ερευνητικό προπολογισμό της Ευρώπης για αμυντικές δαπάνες αφαιρούμε την προοπτική από τις εθνικές βιομηχανίες να χρησιμοποιήσουν από κοινό τις δυνατότητες τους. Τρίτον, αν το συγκρίνουμε αυτό σε σχέση με τους στόχους της Ευρώπης 2020 δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς ε, συμβάλλει η αμυντική έρευνα για τους ε, στόχους της Ευρώπης 2020. Όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, η συμβολή τους ε, είναι μηδενική. Η επένδυση χρημάτων σε έρευνα με μελλοντικά αποτελέσματα που είναι προτιμότερο να επενδύσουμε αυτά τα χρήματα σε καινοτομίε για το μέλλον. Εδώ βλέπω να διαφαίνεται ένα προβλέψιμο δίλημα για όλους μας. Ορίζοντας 2020. Το πολυετές αυτό πλαίσιο δεν θα χρηματοδοτηθεί τόσο άφθονα όσο θα θέλαμε όλοι. Τα κράτη-μέλη ήδη μελετούν το πόσο θα περικόψουν για αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν πιστεύω ότι η έρευνα θα εξαιρεθεί 100% από τις συνέπειες αυτού του αγώνα περικοπών. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες εκεί όπου έχουν την καλύτερη απόδοση. Εκεί όπου υπάρχει καλύτερη προστιθέμενη αξία. Και αυ, αυτός τέτοιος τομέας σίγουρα δεν είναι η αμυντική έρευνα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι εδώ αν ακολουθήσουμε τις συμβουλές σας θα κάνουμε ένα τεράστιο λάθος ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά και θέλω να διατυπώσω, ότι, να δηλώσω σαφώς ότι η ομάδα μου αντιτίθεται σε αυτή την εξέλιξη και ότι θα κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν ώστε να μείνουμε πιστοί στην αρχική συμφωνία που είχαμε και σε αυτή την Επιτροπή στο παρελθόν ότι θα προωθούμε την ε, έρευνα για την ασφάλεια αλλά ότι θα απορρίψουμε την έκκληση τη δική σας για να κινηθούμε προς μια νέα κατεύθυνση χρηματοδότησης της αμυντικής έρευνας ε, και των αμυντικών προμηθειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Λούλη. Ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά τα οποία είπε ήδη ο κύριος Μπίντικ Χόφερ. Θα ήθελα <clears throat> να επανέλθω στο ότι στο κόμμο 809 στο άρθρο 16 πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει στρατιωτική έρευνα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 12. Με παρακολουθείτε, δεν νομίζω. Δηλαδή, στο άρθρο αυτό, αυτό προσπαθεί να εξασφαλιστεί. Το ερώτημα είναι βέβαια πώς αυτό πρόκειται να ε, ε, εφαρμοστεί και ε, θα ήθελα γι' αυτό να διατυπώσω το ερώτημα σχετικά με το πώς το άρθρο αυτό πρέπει να ερμηνευτεί. Το ερμηνεύουμε μήπως διαφορετικά από ότι είναι ο αρχικός του στόχος ε, όσον αφορά ε, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προσπαθούμε να να μην εξάγουμε τεχνολογία η οποία οδηγεί ε, ε, σε τραυματισμούς ανθρώπων. Στο άρθρο 12 λέγεται ότι για την εφαρμογή του ορίζοντα 2020 ε, θα πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχει καταρτήσει η Κομισιόν και ε, θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα προχωρήσουμε διότι η ε, εμπειρία μας απέδειξε ότι σε αυτά, αυτές τις επιτροπές υπάρχουν απλούστατα στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών. Άρα πώς είναι δυνατόν να προγραμματίσουμε κάτι τέτοιο. Έχω άλλη μία ερώτηση σχετικά με τη γραμμή του προϋπολογισμού. Στο κεφάλαιο 6.3 παράγραφος 11 λέγεται ότι για την αναφερόμαστε στην εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και στην άμυνα χωρίς ε, να παραπέμπει κανείς εις ε, τους εξοπλισμούς. Όσον αφορά τις καινοτόμες ε, ε, δραστηριότητες λέγεται ρητός ότι αυτές πρέπει να απευθύνονται μόνο σε πολιτικές δραστηριότητες. Οπότε ε, όπως και ο κύριος Μπίτικ Χόφερ έχουμε διευκρινίσει ορισμένα σημεία και πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ορισμός που αποδίδουμε στην ασφάλεια των πολιτών. Διότι λέγεται σαφώς ή περιγράφεται ότι η κατάσταση των ε, πολιτών στην Ευρώπη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν όταν κοιτάμε τις στρατηγικές ε, κάτι δεν πάει καλά διότι βλέπουμε ότι ιδίω ε, στο κέντρο της Ευρώπης οι πολίτες είναι πιο ασφαλείς από ό,τι ποτέ. Άρα πώς μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά με τη ζωή των γονιών και των ε, ε, παππούδων μας διότι βλέπουμε ε, ότι τώρα υπάρχει μεγαλύτερη ευημερία, λιγότερη υπαρξιακή ανησυχία και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν κάνουμε έρευνα υπέρ της ασφαλείας και όχι να προωθούμε στρατιωτικά προγράμματα διότι εγώ ήμουνα κοινωνική λειτουργός και είδα ε, ε, πώς ήταν η έρευνα, ε, προληπτική έρευνα την οποία κάναμε που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συζητούμε σήμερα και κάτι τέτοιο πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη δηλαδή πώς μπορεί κανείς να προλάβει τη βία να ερευνήσει την πρόληψη της βίας ε, η πολιτική μου ομάδα άρα δεν πρόκειται να στηρίξει αυτή την κατεύθυνση την οποία έχει λάβει η έκθεση την οποία παρουσιάσατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Μπιτικόφερ ήταν πολύ ομός, οπότε μπλάντ όπως είπε. Και θα είμαι και εγώ το ίδιο. Σχετικά με ε, την έκθεση ε, του εισηγητή πρέπει να πω ότι ε, το πνεύμα βασίζεται στις εκθέσεις Ντονζόν και Λίζεκ και συμφωνούμε. Βεβαίως δεν αναφερόμαστε μόνο στη στρατιωτική ασφάλεια διότι σε πολλούς τομείς η ασφάλεια είναι μία πτυχή αλλά όχι μόνο στον τομέα των ε, στρατιωτικό. Και αυτό αληθεύει. Όσον αφορά την ε, τροπολογία 14 ε, εις την γνωμοδότηση λέγεται ο Research and ότι η έρευνα ε, θα πρέπει ε, να ασχοληθεί ουσιαστικά λέγεται ρητός primarily δεν υπάρχει δηλαδή μία μετακίνηση προς ε, έρευνα αμυντική βεβαίως είναι ανόητο να θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν υπάρχει μία αλλαγή προσανατολισμού. Απλούστατα θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα για τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε, παραδείγματος χάρη στις αποστολές μας. Ε, στην ε, ε, εξωτερική δύναμη να υπάρχουν και collateral profits από άλλους τομείς υπέρ των πολιτικών μας αυτό τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο διερευνούμε και θέλουμε να επιτύχουμε. Όχι αποκλειστικά αμυντική έρευνα, αλλά έρευνα τα οποία θα είναι προς όφελος των αποστολών τις οποίες οργανώνουμε. Εάν δηλαδή ε, υπάρχει μία συνεργασία πολιτική ε, μεταξύ των ε, κατασκευαστών ελικοπτέρων η συνεργασία αυτή είναι και πολιτική και στρατιωτική διότι προωθούμε την υψηλή τεχνολογία και θα υπάρξουν αποτελέσματα και για την βελτίωση ενός ελικοπτέρου το οποίο χρησιμοποιούμε σε στρατιωτικές αποστολές. Απλούστατα λοιπόν δεν πρέπει να προσπαθήσουμε τεχνητά να αποφύγουμε να υπάρχει μία προώθηση στον στρατιωτικό τομέα ενός αποτελέσματος ερεύνης στον πολιτικό τομέα διότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο θαραλέοι στον τομέα της αμήνης και να θέτουμε στόχους. Άρα υπάρχει μία προστιθέμενη αξία στον τομέα της ερεύνης και στο στρατιωτικό τομέα για τις αποστολές όπως τόνισα διότι παραδείγματος ε, χάρη τα drones, αυτά ε, τα ε, οχήματα τα οποία όπου δεν υπάρχει άνθρωπος που να τα οδηγεί είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το, τις κλιματολογικές αλλαγές πηγαίνοντας πάνω από το δάσος του ε, Αμαζονίου να έχουμε αποτελέσματα δηλαδή της ερεύνης με μη επανδρομένα αεροσκάφη και ε, αυτά να μπορούμε ε, να τα χρησιμοποιήσουμε σε πολλά επίπεδα δεν είναι κάτι κακό οι αποστολές που αποφασίζονται από τις κυβερνήσεις είναι ηλιμένες αποφάσεις και έχουν επιπτώσει σε διάφορα επίπεδα ακόμη και στο στρατιωτικό όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα της ερεύνης. Δεν αλλάζουμε εστιασμό του προγράμματος, απλούστατα μπορούμε πολιτικά να πούμε ότι χάρη σε την στήριξή μας ή ε, την έρευνα ε, και την αριστεία έχουμε επιτύχει αποτελέσματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην αμυντική μας πολιτική. Εξού και στηρίζω την ε, οπτική γωνία του εισηγητή και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο χαλαρά και να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι με αυτά τα οποία λέγονται εδώ μπορούμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια από τους εθνικούς αμυντικούς προπολογισμούς. Η κυρία Λόζινγκ. Χωρίς μικρόφωνο. Εδώ βεβαίως είμαστε μία ε, υποεπιτροπή της Επιτροπής Εξωτερικών. Γι' αυτό το λόγο ε, ακόμη και αν έχω διαφορετικές απόψεις και δεν είναι κάτι που θα, ε, θα αναφέρω εδώ, μπορούμε να έχουμε διαφορετική άποψη για την εξωτερική πολιτική. Αλλά τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται στις συζητήσεις έχουν και αποτελέσματα εσωτερικής πολιτικής σε ολόκληρο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εξού και σχετικά με την έρευνα αυτή πρέπει να αναρωτηθούμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για άμυνα. Γνωρίζω την έκθεση των Ζων και τις άλλες διότι στις εκθέσεις αυτές η οπτική γωνία δεν στηρίζεται. Εμείς θεωρούμε ότι το βασικότερο στοιχείο είναι η ασφάλεια και η ευημερία των ανθρώπων στην Ευρώπη και στον κόσμο πρέπει να δούμε με ποιον, ε, ε, ε, σε τι αποβλέπει η έρευνα την οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή τι, πώς θα επηρεάσει τα δικαιώματα του πολίτη, τη δημοκρατική εξέλιξη, τι σκοπούς επιζητεί. Αυτό που είπε ο κύριος Γκάλερ με ανησυχεί πολύ, δηλαδή στις επόμενες διαδηλώσεις θα μπορεί να χρησιμοποιήσει καλής μη επανδρομένα αεροσκάφη ε, ε, διότι εσείς αναφέρατε ορισμένα παραδείγματα εγώ όμως σκέφτηκα ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι και πρέπει να θέσουμε τα αιτιολογημένα μας ερωτήματα και να δούμε σχετικά με τον προϋπολογισμό τι μέλη όταν μιλάμε για χρήση του κονδυλίου 6 του προϋπολογισμού για τις καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αμυντική έρευνα και πώς κατατάσσονται. Ευχαριστώ. Mr. Luhan. Yeah. Ähm, Ευχαριστώ. Υπήρξαν ορισμένες ιδέες τις οποίες παρουσίασε ο κύριος Μπίτι Κόφερ και η κυρία Λέζινγκ ε, και τα σεύχομαι πάρα πολύ, ε, τα συμφωνώ. Με συγχωρείτε λέει ο μιλητής που σας είπα κυρία Λούλινγκ και όχι κυρία Λέζινγκ. Σχετικά ε, με ε, τα σχόλια. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσει η έρευνα και η ανάπτυξη σε τομείς σαν αυτόν που μας απασχολεί. Τώρα, εάν θα υπάρξει ε, υψηλότερη ή λιγότερη επίπτωση στην οικονομική εξέλιξη είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν, κατά τη γνώμη μου, στον τομέα αυτό σήμερα να μείνουμε πίσω. Ιδίως διότι άλλες χώρες, άλλες στρατιωτικές δυνάμεις επενδύουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε αυτό τον τομέα όπως η Αμερική, η Κίνα, η Ιαπωνία και πολλές άλλες μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο την οικονομική πτυχή και πολύ σωστά ε, ο κύριος Γκάλερ είπε ότι ουσιαστικά τα ποσά είναι ελάχιστα αν τα συγκρίνει κανείς με άλλα ποσά του κοινοτικού προπολογισμού όσον αφορά την ασφάλεια. Στον τομέα αυτό δεν πρέπει μόνο να εστιαστούμε στην ανάπτυξη οπλισμών ε, όταν μιλούμε για research and development, για έρευνα και αναπτυξή, αλλά να εξετάσουμε και την πτυχή της ασφάλειας και να δούμε τι γίνεται εκεί. Μήπως χρειάζομαστε ε, δραστηριότητες έρευνας και αναπτύξεως ή όχι. Κατά τη γνώμη μου τις χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ, διότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις ε, δεν είναι τόσο πίσω στο παρελθόν οπότε όπως είπατε και εσείς η ίδια κυρία Λέζινγκ η πρόληψη είναι καλύτερη από την ε, επέμβαση εκ των υστέρων και στο πνεύμα αυτό θα έπρεπε να αποδώσουμε στον τομέα αυτό την σημασία που του πρέπει και επαναλαμβάνω ιδίω εφόσον τα ποσά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Έχετε βέβαια δίκιο όταν λέτε ότι εδώ θα ε, δεσμεύσουμε ένα ποσό και πόσο θα το κατατάξουμε. Δηλαδή ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες θα περιληφθούν στο κονδύλι αυτό. Είναι κάτι προς συζήτηση. Πρώτα πρέπει να συζητήσουμε τι θέλουμε να ερευνήσουμε ή πρώτα πρέπει να πούμε ότι θα δεσμεύσουμε ένα αλφα ποσόν για αυτές τις δραστηριότητα και στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου του προϋπολογισμού θα προβούμε σε μία συζήτηση όσο προς τους στόχους. Είναι κάτι που μπορούμε να διευκρινίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ε, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Εγώ βλέπω ότι στην Επιτροπή, την Περιφερειακή Επιτροπή ε, που τα ποσά είναι τεράστια ε, γίνεται η ίδια διαδικασία. Λέμε ότι θα δεσμεύσουμε αυτά τα ποσά για την συνοχή και μετά βλέπουμε πώς θα κατακαιρματιστούν. Είναι ουσιαστικά θέματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσουμε καταρχήν επί γενικής βάσεως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και οικονομικά ωφέλη, τα οποία θα αποκομίσουμε και ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ευελιξία σχετικά με τον τομέα της ασφάλειας και της αμήνης. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Πιστεύω ότι πρέπει να στηριχτεί. Και αντιλέγω τον κύριο Μπίτικόφερ και την κυρία Λόιζινγκ, διότι εγώ δεν νομίζω ότι ζούμε στην πλέον ασφαλή κοινωνία σήμερα. Πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κίνδυνοι. Κίνδυνοι οι οποίοι δεν υπήρχαν πριν από την τεχνολογική εποχή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίως χρειάζεται να έχει αρμοδιότητες στρατιωτικές ε, η Ευρώπη. Δεν λέω το αντίθετο. Λέω όμως ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ειλικρινά σύμφωνα με την αρχή του να τα βάλουμε όλα από κοινού και να τα μοιραστούμε όλα μεταξύ μας. Ας κάνουμε όμως μία διαφοροποίηση. Τι θα κάνουμε με τον προϋπολογισμό για την έρευνα του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ε, ήρθα σε αυτή την επιτροπή μου είπε και ο κύριο έχουμε μία συμφωνία, χρηματοδοτούμε την έρευνα για μη στρατιωτικού σκοπούς, αλλά όχι για στρατιωτικούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξιολογήθηκε, εκτιμήθηκε και αποδεικνύεται ότι δύο, τρία, των, δύο τρίτα των συνολικών δαπανών πήγανε σε μία μόνο ε, γαλλική εταιρεία, την Ταλής. Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ αποδοτική. απέδωσαν τα ερευνητικά τους προγράμματα, έτσι όπως οριζόταν στο παρελθόν. Δεν είμαι θεροβάμων, ούτε αισιόδοξο τόσο πολύ, για να πιστέψω ότι αν επιτρέψουμε έρευνα σε προγράμματα που αφορούν εφαρμογές μη στρατιωτικές θα ωφελήσουμε τους στρατιωτικούς. Αλλά εδώ πρέπει να πω ότι εδώ έχουμε, ε, δεν έχουμε ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή. Αυτό προσπαθώ να πω και δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Στην αιτιολόγηση λέει ο εισηγητής ο εισηγητής θεωρεί ότι το άρθρο 16.2 είναι ιδιαίτερα προβληματικό, δεδομένου ότι αναφέρει ότι οι δραστηριότητες καινοτομία και έρευνα στα πλαίσια του Horizon 2020 πρέπει έχουν αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι, δεν, ότι αποκλείεται οποιαδήποτε στρατιωτική φύση έρευνα από το πρόγραμμα. Αυτό θέτει σε αμφισβήτηση και νομίζω ότι αυτό κύριε Γκάλη, συνάδει με αυτό το οποίο είπατε, ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι μη στρατιωτική, εμπορική στόχη, και όταν χρησιμοποιείτε τον όρο κυρίω primarily, σημαίνει ότι έρχεται και κάτι μετά, κατά δεύτερον. Και αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά. Μέχρι τώρα επιτρέπαμε μόνο, και αυτό είναι τώρα το νέο ερευνητικό πλαίσιο το πολιετές, μέχρι τώρα επιτρέπαμε σε αυτά τα πλαίσια να γίνεται έρευνα εστιασμένη σε μη στρατιωτικού στόχου παρά το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως και σε διπλή εφαρμογή, σε διοική εφαρμογή. Έτσι λοιπόν μπαίνει το παραθυράκι το στρατιωτικό τομέα και αυτό είναι διαφορετικό. Πράγμα το οποίο δεν συνάδει με αυτό που είχαμε ψηφίσει προηγούμενε εκθέσει. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ την διατύπωση και την διατύπωση σε όλες τις γλώσσες. Αλλά αυτή η διατύπωση ξεπερνάει την κόκκινη γραμμή. Ο κύριος Λουχάν μίλησε για την ε, κυβερνοέρευνα. Αυτό δεν είναι θέμα αποκλειστικά στρατιωτικό. Πρόκειται για μία πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλοι οι, οι τομείς και η τρομοκρατία που είναι η χειρότερη κυβερνοεπίθεση στον κόμμα μας είναι κάτι το οποίο επιτρέπουν και δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις δύο χωρών με τις οποίες έχουμε και στενή σχέση. Όταν λοιπόν βγει στην επιφάνεια ένα τέτοιο είδος ε, μικρόβιο, ενα τέτοιος ιός, κάποια στιγμή θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Εντάξει, ωραία στην έρευνα, στην αντίσταση κατά των εγκλημάτων στον ε, κυβερνοχώρο, αλλά να μην ξεπεράσουμε και την κόκκινη γραμμή, είπαμε, μεταξύ αυτών που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασφάλειας και της άμυνας και των δαπανών τους για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Σε κάποια από τα έγγραφα που κυκλοφορούν, είδα ότι κάποιοι συνάδελφοι σκέπτονται ακόμη και να χρηματοδοτήσουν και κάποιες δημόσιες συμβάσεις κάπου σε κάποιες χώρες. Πράγμα το οποίο διαφωνεί με τη γραμμή που ακολουθούμε. Και επιμένω στο επιχείρημά μου. Θα πρέπει να πάρουμε μια πολύ ενσυνείδητη απόφαση. Θέλουμε να εμείνουμε σε αυτά που κάναμε μέχρι τώρα ή θέλουμε να ανοίξουμε νέα πόρτα, μεγάλη πόρτα, ώστε να μπει και η στρατιωτική έρευνα ε, από τα κονδύλια του κοινοτικού προσμού. Θέλουμε να γίνει έρευνα περαιτέρω για τα μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη. Ναι, αλλά Εμεί με τα δικά μας κοινωτικά κονδύλια να τα χρηματοδοτήσουμε. Όχι κύριε Γκάλερ. Τώρα, σε σχέση με το τελευταίο επιχείρημα του κυρίου Λουχάν, είπατε επιπτώσεις στην ε, οικονομική ανάπτυξη Δεν νομίζω ότι έτσι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χρήματα των ε, Ευρωπαίων φορολογουμένων. Όντως εστιαζόμαστε σε δραστηριότητες έρευνας. Είναι μια συμφωνημένη πολιτική μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Όντως, χρηματοδοτούμε αυτές τις δραστηριότητες για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ε, της ε, οικονομικής ε, ανάπτυξης. Τώρα, Uh, research contributes or not. No, it, it's not. Τώρα, το θέμα αυτό, το πού θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα όσον αφορά το ποσό. Σωστά. Το ποσό το οποίο μπορούμε να παράσχουμε δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης χρηματοδοτώντας ε, κάποιες δραστηριότητες στον κοινωτικό προβλησμό. Συμφωνώ. Πλην όμως πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να δούμε ότι κάποια συμφέροντα κοιτούν επίμονα τις τσέπες μας και πώς θα τους χρηματοδοτήσουμε και βεβαίως η ευρωπαϊκή αμυντική ε, βιομηχανία θέλει χρήματα και θα ήθελε να κάνει κάποιες ρυθμίσεις και συμφωνίες για να προωθήσει τις δαπάνες για στρατιωτικούς λόγους. Διότι τελικά έχουν γίνει και μεγάλοι γραφειοκράτες. Είναι λυπηρό αυτό. Πιστεύω ότι η δική του προσέγγιση επίσης θα πρέπει να είναι κάπως διαφορετική. Και πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε ό,τι διαθέτουμε από κοινού και να το μοιραστούμε μεταξύ μας. Δεν λέω ότι η έρευνα στον τομέα το στρατιωτικό δεν είναι κάτι το σωστό. Λέω όμως ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομιμοποιούμεθα να προχωρήσουμε σε αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Θα λάβω υπόψη τις ε, έντονες αντιρρήσεις που ακούγονται εδώ από τους συναδέλφους και ελπίζουμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνουμε μια συνεδρία σχεδόν και θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο προσέγγισης του ζητήματος καθώς και τη σωστή διατύπωση ώστε να γίνει πιο αποδεκτό και να μην γύρει τις αντιρρήσεις που ακούσαμε σήμερα εδώ. Επίσης Ας έχουμε υπόψη μας ότι αυτή είναι μια προσπάθεια να συμπεριλάβουμε κάτι σε σχέση με την άμυνα και τη σχετική έρευνα στο ορίζον 2020. Σε αυτό το εγχείρημα η γνωμοδότηση μας λοιπόν προσπαθεί να προσθέσει κάτι από τη δική μας άποψη ως Υποεπιτροπής Άμυνας αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί ως ένα εγχείρημα να συμπεριληφθεί κάτι στο Horizon 2020. Θα λάβουμε υπόψη φυσικά τα σχόλιά σας, αλλά δυστυχώς θα χρειαστεί να συνεχίσουμε αφού ακούσουμε τους ομιλητές που βρίσκονται εδώ, να καλέσουμε τον Ναύαρχο να λάβει το λόγο. Καλούμε λοιπόν τον κύριο στρατηγό να λάβει το λόγο. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας ε, σε σχέση με τη συζήτηση που μόλις έλαβε χώρα. Προτείνω η Επιτροπή και ε, η Υπηρεσία να λάβουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των συναδέλφων μας μετά από την ακρόαση του στρατηγού Σιρέν. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε για άλλη μια φορά μαζί μας τακτικά ανταλλάσσουμε απόψεις και σήμερα η ακρόαση αυτή θα αφορά κυρίως τις τρέχουσες στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις με φυσικά τις δύο ε, εμβληματικές ε, επιχειρήσεις Αταλάντα και UTM ε, Σομαλίας όσον αφορά το κέρας της Αφρικής και τη συνέχιση της ε, αποστολής Ανθέας στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Τρεις λοιπόν νέες αποστολές ε, έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Πρόκειται για μη στρατιωτικέ, αλλά μία ιδιαίτερωση καπνεστόρ που αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και υποδομών στα κράτη του κεράτος της Αφρικής για την καταπολέμηση της πειρατείας περιέχει μία στρατιωτική συνιστόσα και ένας ε, τέος ε, Γάλλος Ναύαρχος ε, βρίσκεται επικεφαλής αυτής της αποστολής και έτσι μπορεί να μας πει ίσως δύο λόγια για αυτή την αποστολή. Πέραν των επιχειρήσεων θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας όσον αφορά την ενεργοποίηση του Op Center που ε, οδήγησε σε πολλές συζητήσει πέρυσι αυτή η απόφαση για την ενίσχυση των διαφόρων επιχειρήσεών μας στο κέρας της Αφρικής. Ε, αν έχετε κάποιες απόψεις ε, να μοιραστείτε μαζί μας επί του θέματος θα ήταν πρόσδεκτες. Και τέλος όσον αφορά τις ικανότητες που βρισκόμαστε κατά την άποψή σας στο πλαίσιο του pooling and sharing, της συγκέντρωσης πόρων και της κοινής χρήσης, πώς εσείς θεωρείται ότι ήταν τα συμπεράσματα της ε, Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Σικάγο και η ενεργοποίηση του pooling and sharing σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι θέματα που μας ε, αφορούν πρωτίστως. Ε, αυτά σας προτείνω να είναι η θεματολογία μας σήμερα το πρωί. Σας έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και για αυτή την... αυτό το πλάνο. Θα τα καλύψω όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, εκτιμώ ιδιαίτερα την προσκλήσή σα για μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σα. Έχουν περάσει δύο χρόνια από την τελευταία φορά είχα πολλές επαφές με πολλούς από εσάς κατά την προετοιμασία των δικών σας εκθέσεων για την κοινή πολιτική και των εκθέσεων σε σχέση με τις αμυντικούς προπολογισμού πριν δύο χρόνια έδωσα την άποψή μου για το CSDP και τη στρατιωτική διάσταση περίπου έξι μήνες μετά από την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας μίλησα για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιτροπής ε, για τη διαδικασία υλοποίηση και ειδικότερα για τη μόλις τότε συμφωνηθήσεις προτεραιότητες ε, για τη στρατιωτική επιτροπή μου. Επίσης σχολίασα για τις ε, ενεξελίξει επιχειρήσεις και επίσης ε, συζήτησα για τις προ... Ε, προχωμένες προκλήσεις και δεδομένων και των περικοπών του προπολογισμού. Σήμερα ξεκινάω με μια σύντομη εισαγωγή ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Κοιτώντας τα προηγούμενα διδάγματα που έλαβα ως πρόεδρος, θα κοιτάξω τα πράγματα αναδρομικά αλλά και με ένα μάτι προς το μέλλον. Αντιλαμβάνομαι ότι μία από τις ε, σπάνιες ευκαιρίες που έχω να εκφράσω και τη δική μου προσωπική άποψη είναι τώρα, κοντά στο τέλος της θητείας μου ως Θα ξεκινήσω με σχόλια για την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας από την άποψη της Στρατιωτικής Επιτροπής. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση, σας δηλώνω αμέσως ότι είμαι περισσότερο πεπισμένος από ποτέ για την αξία και την αναγκαιότητα πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ των κράτων μέλων στο στρατιωτικό τομέα. ξεκινώντα για μια ενισχυμένη κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνα στην Ευρώπη, συγχωνεύοντα ξεχωριστού όργανα και καθιερώνοντας διαφορετικές και με καθιερωμένε διαφορετικέ προτεραιότητε και πρότυπα, όλα αυτά χρειάζονται πολλή δουλειά στις Βρυξέλλες τα τελευταία δύο χρόνια. Είχα θεωρήσει ότι θα ήταν πιο σύντομη η διαδικασία, παρότι αντιλαμβάνομαι τι δυσκολίε και τι προκλήσει λόγω των διαφορετικών καθιερωμένων οργανισμών και σωμάτων που προσπαθούμε να συγχωνεύσουμε σε ένα ενίο πλαίσιο. στη Στρατιωτική Επιτροπή το να μοιραστούμε τις 27 διαφορετικές απόψεις των 27 ε, διαφορετικών κρατών μελών σε αυτή τη διαδικασία αντιλήφθηκα πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε την υπομονή παρότι η υπομονή δεν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά, από τις πιο χαρακτηριστικές μου ιδιότητες, αλλά η συνεργασία σε διάφορους τομείς θα πρέπει να ε, έχει το χρόνο που χρειάζεται. Προσωπικά προσπαθώ να κάνω συζητήσεις σε ζητήματα που θεωρούνται ε, περιφερειακά προς την ίδια την ειρηνευτική διαδικασία. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πιεστούν περισσότερα καθώς ε, τώρα λαμβάνει πλήρη ταχύτητα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης για αρκετό καιρό ε, χάσαμε κάποιες από τις αλλαγές που είχε που... αλλά τώρα ελπίζουμε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να λειτουργήσει προενεργά Κοιτώντας τα επιτεύγματα μας από το 2009 πρέπει να διατρούμε στο μυαλό μα διαφορου παράγοντε. Μπορούμε να πούμε ότι οι προκλήσει ήταν πολύ μεγαλύτερε από ό,τι αναμέναμε πριν από δύο χρόνια. Η περίοδος ε, προετοιμασίας ε, συνέπεσε με μία από τις πιο τραχώδεις εποχές ε, στον κόσμο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ψυχρό πόλεμο. Η αλλαγή του πόλου εξουσίας ε, ισχύω από την Ευρώπη προς την Ασία, η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επαναστατικές αλλαγές στη Βόρεια Αφρική, όλα αυτά ε, έθεσαν νέα δύσκολα καθήκοντα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά την ανάπτυξη η ανάπτυξη των διαδικασιών για τη CSDP δεν ήταν προτεραιότητα στα κράτη-μέλη. Η δική μας άποψη είναι παγκόσμια, καθολική, αλλά η πρόσφατη εμπειρία μας θυμίζει ότι η σταθερότητα του στενού μας περιβάλλοντος δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Παρότι η αποστολή εκπαίδευση στην Ουγγάντα ξεκίνησε το 2010, καμία νέα επιχείρηση CSDP δεν έχει ξεκινήσει από το 2008. Παρότι μειώθηκε ο αριθμός των στρατευμάτων, ήταν ευκολότερη η διαμόρφωση πολιτικών φιλοδοξιών ε, που να ε, σχετίζονται με στρατιωτικές δεσμεύσεις. Τελικά αυτό είναι ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Είναι εύκολο στα λόγια, δύσκολο στις πράξεις. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι η στρατιωτική διάσταση του CSDP χρειάζεται πολιτική προσοχή και προτεραιότητα. Είναι δύσκολο να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά τα κράτη-μέλη έχουν ένα σύνολο δυνάμων και ό,τι κάνουν στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συνδέονται στενά. Έχουμε τις περιπτώσεις του Αφγανιστάν, του Κωσυφοπεδίου, της Λιβύης, που κατέστησαν δύσκολη τη διαχείριση και την οικονομική στήριξη άλλων δεσμεύσεων. Αξίζει να θυμόμαστε ότι τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει με περισσότερους από 30.000 στρατιώτες σε συνεχή βάση. Οι στόχοι είναι παράλληλοι με τους στόχους της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφαλείας. Απομένει να δούμε πώς θα οριστούν οι προτεραιότητες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ όταν τα στρατεύματα στο Αφγανιστάν θα έχουν μειωθεί σημαντικά περίπου στο 2014. Από την άλλη πλευρά, εγώ αντιλαμβανόμαι ότι το πολιτικό ενδιαφέρον για... είναι περιορισμένο για νέες επιχειρήσεις. Μια νέα προσέγγιση του επιμερισμού φόρτου διατλαντικά ε, με έναν πιο ισχυρό ρόλο της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ και το γεγονός ότι όλα τα κράτη-μέλη σήμερα πλέον έχουν ενταχθεί στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ θα αυξήσει το ενδιαφέρον ώστε το ΝΑΤΟ να είναι το πλαίσιο για τη διαχείριση των πολιτικών κρίσεων όταν αυτό είναι πολιτικά δυνατό. Η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας είναι η, δυνατότητα χρήση όλων των μέσων, στρατιωτικών και μη, με αποτελεσματικό και ολοκληρωτικό τρόπο περισσότερο από ποτέ. Είμαι πεπισμένο ότι η επιτυχή ανάπτυξη και χρήση τη ε, κοινή προσέγγιση βασίστη συνθήκη τη της θα αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία τη κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνα Με αυτή την προσέγγιση υπάρχει και μια σημαντική στρατιωτική διάσταση το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή για το κέρας της Αφρικής ε, δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος το πρόγραμμα Νέστορ, το οποίο τώρα έχει ενσωματωθεί και στην αποστόλη εκπαίδευση και στην επιχείρηση Αταλάντα στο πλαίσιο της όλης στρατηγικής για το κέρας της Αφρικής. Επαναλαμβάνομαι, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η πρώτη δοκιμασία της πραγματικής ολοκληρωμένης προσέγγισης. Αναμένουμε ακόμα τη χρήση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού, αλλά καλή αργά παραποτέ είμαι πεπισμένος ότι σήμερα βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, διασυνδέοντας τις διάφορες δραστηριότητές μας εντός και εκτός Ομαλίας. Η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαδραματίσει ρόλο για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας έχει προληπτικά ανταποκριθεί διατυπώνοντας τις στρατηγικές της προτεραιότητες πριν δύο χρόνια και έτσι έδωσε προτεραιότητα στην υποστήριξη και την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας και μάλιστα στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η υποστήριξή της Στρατιωτικής Επιτροπής εκφράστηκε στις πέντε στρατηγικές προτεραιότητε που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις ιδέες και τις προθέσεις της συνθήκη της Λισαβόνας πρώτα απ' όλα βασικές ε, ενεξελίξει επιχειρήσει, δεύτερον μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιόπιστη ανέφερα τη στρατηγική του στο κέρας της Αφρικής, στρατηγικές ε, συνεργασίες, ΝΑΤΟ, Ηνωμένα Έθνη, μεμονωμένα κράτη-μέλη και η ανάπτυξη δυνατοτήτων και υποδομών ικανοτήτων και τέλος άμεση υποστήριξη για την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτές είναι οι 4-5 προτεραιότητες με τις οποίες ασχολούμαστε σε καθημερινή βάση στη Στρατιωτική Επιτροπή. Τίποτα άλλο. Η Στρατιωτική Επιτροπή έχει αποτελέσει καταλήτη για μια ρεαλιστική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό απεικονίστε στα διάφορα θέματα που έχουμε στις σημερινές διατάξεις μας στις τελευταίες συνεδριάσεις ε, επικεφαλής ε, άμυνας και ε, στην αρχή έχουμε τη συγκέντρωση πόρων και την κοινή χρήση και την πρόληψη σειράξεων. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί και στο κέρας της Αφρικής οι στρατηγικέ προτεραιότητε υπήρξαν χρήσιμε όχι μόνο για το δικό μας έργο, αλλά και για άλλες πτυχές ε, της κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας δεδομένου ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η φάση υλοποίηση. έχουν προσαρμοστεί οι προτεραιότητε αντίστοιχα. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω ώστε να συζητήσουμε για το μέλλον όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτή είναι η δεύτερη στρατηγική μας προτεραιότητα. Έχω επισκεφθεί σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη. Μέσω των διμερών μου συζητήσεων απέκτησα μια πολύ καλή εικόνα των διαφόρων ε, καταστάσεων σχεδιασμού σε όλες τις χώρες όσον αφορά την άμυνα, οι τεράστιες περικοπές, οι τεράστιες αυξήσεις των δαπανών που σχετίζονται με τις νέες γενιές εξοπλισμών, η μεταβόλη του φόρτου και τα υψηλά κόστη των διαρκών επιχειρήσεων δημιουργούν διλήμματα σχεδιασμού. Διαρκώς τους ζητείτε να κάνουν περισσότερα με λιγότερους σπόρες. Τα πολλά κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα μέσα στα επόμενα χρόνια. Οι πρόσφατες δημοσιονομικές περικοπές έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα και έχουν κάνει τα προβλήματα πιο ορατά. Αλλά υπογραμμίζω κάτι που είναι ανεξάρτητο από αυτές τις ε, περικοπές. Τα βασικά προβλήματα, ανεξάρτητα από αυτές τις περικοπές, είναι ότι οι άμυνες κοστίζουν όλο και περισσότερο και ότι κάνουμε ελάχιστες προσπάθειες για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ότι, οι αποφάσεις που λαμβάνουν, και ότι έχουμε αποφάσεις που λαμβάνονται σε 27 εθνικά πλαίσια. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα περικοπών και λιτότητας, είναι και το πώς κάνουμε τη δουλειά μας σε ένα ενώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχουμε επανάληψη εργασιών, επικαλύψεις και θα έλεγα ότι το κύριο μας πρόβλημα δεν είναι ότι ξοδεύουμε πολύ λίγο για την άμενα. Εξάλλου τα 27 κράτη-μέλη ξοδεύουν 200 δις ευρώ το χρόνο για την άμυνα. Αυτό είναι μόλις το 1 τρίτο των δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα, αλλά ισούται περίπου με το άθροισμα της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Σαουδικής Αραβίας, πέντε χώρες οι οποίες, των οποίων οι αμυντικές δαπάνες αθροίζονται και ισούνται με την με τις ευρωπαϊκές δαπάνες. Πρέπει λοιπόν να, με κριτικό πνεύμα να δούμε πώς θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποδοτικοί στις δαπάνες μας. Πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες για καλύτερες ικανότητες σε περίπτωση που μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα τις προσπαθίες μας. Φυσικά εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω τα ζητήματα κυριαρχίας. Η κυριαρχία φυσικά, η εθνική κυριαρχία είναι ένα από τα κύρια ζητήματα εδώ όταν λαμβάνει αποφα... όταν λαμβάνεται αποφάσεις οποιοδήποτε κράτος μέλος αλλά είναι σαφές κατά την απόψη μου ότι αν εμείς τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούσαμε λιγότερα πιο ευρωπαϊκή πτυχή, ε, ε, η εικόνα θα ήταν τελείως διαφορετική. Ε, γνωρίζουμε τις πρωτοβούλες του 2010 από τους Υπουργούς Άμυνα που έθεσαν τα θεμέλια για καλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω μιας πιο στενής εργασίας μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων. Το pooling and sharing έχει γίνει λέξη κλειδί για τις προσπάθειές μας. Μας στηρίζει η EDA, η Στρατιωτική Επιτροπή και η EDA, η Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, συνεργάζονται στένα. Παρόμοιες προσπάθειες ε, γίνονται και στο ΝΑΤΟ. Στόχοι είναι οι ίδιοι και οι προσπάθειές μας άλλοι ε, υποστηρίζονται και είναι συμπληρωματικές. Έχουμε επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κατάλογο υποσχόμενων προγραμμάτων. Ορισμένα από αυτά έχουν αρχίσει να αποδίδουν ικανότητες και υποδομές. Θα ήθελα ωστόσο να είμαι πολύ σαφής. Αυτό είναι μόνο το τέλο τη αρχή. Έχουμε τη μεθοδολογία, αλλά αν τα κράτη-μέλη θέλουν πραγματικά να αντιμετωπίσουν τι συνέπειε των άμεσων και μακροπρόθεσμων οικονομικών πραγματικότητων αυτή η συνένωση και κοινή χρήση το pooling and sharing θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Τι μπορεί να μας προσφέρει το pooling and sharing χονδρικά. Τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια σε σύγκριση με τις περικοπές του προϋπολογισμού. Η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από, ότι, από τότε που ξεκινήσαμε. Αλλά διαβάσαμε καλά, έχουμε μια μεθοδολογία και με αυτόν τον τρόπο θα φέρουμε το pooling and sharing σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής και στρατιωτικής νοοτροπίας. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν μπορούμε πλέον να κρυβόμαστε πίσω από γενικολογίε όπως ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα βάσει μια σταθερής κοινή βούλησης να ε, παρακάμψουμε τα, τους εθνικούς φραγμούς και εάν καταφέρουμε να συνεχίσουμε με μια πολιτική προσπάθεια και εγώ βλέπω θετικά μηνύματα ο πρόεδρος Βαν Ρομπόι δήλωσε στο Σύνοδο Κορυφής του Σικάγο ότι έχουμε μια προορετική ε, προσέγγιση ενώπιον κρατών μελών κατέστησε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται σε συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης της δυνατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρά ώστε να, αναλάβει ένα πιο σημαντικό ρόλο ασφαλείας στη γειτονία της και πέραν αυτής. Αυτό υπογραμμίζεται από την πρόσφατη απόφαση συμπερίληψης της άμυνας και της ασφάλειας στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του επόμενου έτους. Και έτσι το ζήτημα ε, ε, γίνεται στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο στους αρχηγούς κρατών. Βλέπω επίσης θετικά σημάδια ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανήσυχεί για τον κατακαιρματισμό της τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη. Έχει δημιουργήσει πρόσφατα μία Task Force Defense για την άμυνα και αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι ενισχύεται η κατανόηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ας μην ξεχνάμε τέλος ότι το ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο ζήτημα εξοικονόμησης χρημάτων, είναι το να διατηρήσουμε τη στρατιωτική μας σπουδαιότητα, αυξάνοντας τη στρατιωτική μας αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε, στρατηγέ μου. είδα ότι θα αποχωρήσετε το φθινόπωρο τα καθήκοντα σας πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε πιο ελεύθερα ίσως να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις του τι είναι και τι πρέπει να γίνει. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε και κυρίως αυτή, αυτό που μας είπατε όσον αφορά τις ικανότητες στο τέλος. Υπενθυμίσατε ότι δεν είναι τόσο θέμα μέσων, έχουν τα μέσα οι Ευρωπαίοι, ακόμη και τα κονδύλια, αλλά ίσως ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα συντονίζουμε τα μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε, διότι εάν ο, τα κονδύλια που δίδει ο προϋπολογισμός των 27 κρατών για την άμυνα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δίνουν οι ΙΠΑ, βρισκόμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι άλλες αναδυόμενες χώρες και δυνάμεις και θα πρέπει να δούμε αν θέσουμε από κοινού όλες τις προσπάθειες θα μπορέσουμε να έχουμε βαρύνουσα θέση και αυτό θα ήταν βεβαίως καλύτερο από το να κάνει ο καθένας στη γωνιά του μόνος του κάποιες προσπάθειες που δεν είναι και τόσο αποδοτικές. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, υπενθυμίσατε και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε από άποψη στρατηγική στο Κοινοβούλιο και πέραν της δικής μας υποεπιτροπής είναι το θέμα της στρατιωτικής διάστησης της ΚΕΠΑ. Το γεγονός ότι μετά την Αταλάντα το 2008 δεν έγινε καμία μεγάλη εμβέλειας επιχείρηση τι καταδεικνύει ότι ίσως δεν υπάρχει μεγάλων ενδιαφέρον εκ μέρους των κρατών μελών, αλλά και μετά την συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές. Δεν ε, λείπουν βεβαίως τα τελευταία χρόνια οι προκλήσεις, ας σκεφτούμε τι γίνεται στο Κάφσασο, στο Σαχέλ, στο κέρας τη Αφρικής. Υπάρχουν κοντά στα σύνορά μας διάφορες ζώνες ανασφαλής ας σκεφτούμε τη Λιβύη. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί, όχι μόνο εκ μέρους των κρατών μελών, αλλά και εκ μέρους των Βρυξελών, για το να προστρέξουμε στο στρατιωτικό σκέλος αυτό της ΚΕΠΑ. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό το πρόβλημα, αν είναι θέμα πιο μακροπρόθεσμης ε, στρατηγικής. Μας έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας ε, φιλόδοξους ε, στόχους και μέσα, τους υπενθυμίσατε. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των ε, κονδυλίων του κοινωτικού προϋπολογισμού και πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει μεγάλη όρεξη να μπουν σε αυτό το δρόμο πολλές χώρες. Το παράδειγμα που δώσετε για το τη Αφρικής είναι ένα παράδειγμα επιτυχές, παρά το γεγονός ότι μετά από την ανάπτυξη κάποιων αποστολών βλέπουμε με ικανοποίηση ε, ποια είναι η σημασία της. Και τώρα βλέπουμε ότι διαθέτουμε αρκετά μέτρα αποδοτικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια γεγονότα και όχι μόνο την πειρατεία, παρά το γεγονός ότι είναι ε, θεαματικό αυτό που συμβαίνει με την πειρατεία, θα έλεγα. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερε ερωτήσεις να κάνω. Ήθελα απλώ να κάνω αυτά τα παρατηρήσεις και αυτά τα σχόλια. Ίσως μια πιο συγκεκριμένη όμως ερώτηση για την Αταλάντη, αν έχετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ευνοϊκές οι κλιματικές ε, συνθήκες και για τους πειρατές, αλλά έχει καταγραφεί στατιστικά αρκετά σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό της ε, εκρίζωσης των επιθέσεων και των καταλήψεων πλοίων. Έχετε μας κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς. Επίσης, Χθε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων συζητήσαμε το θέμα της επέκτασης της εντολής που έχει δοθεί στην Αταλάντη. Κάποιες πολιτικές ομάδες, κάποιοι συνάδελφοι εξέφρασαν ενδιασμούς και στο μέλλον, στο αμέσο μέλλον, πώς βλέπετε εσείς αυτή την προσφυγή σε διάφορες επίγειες επιχειρήσεις πρέπει να συστηματοποιηθούν, ανταποκρίνονται σε ανάγκες των επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι κάποιες χώρες που συμμετέχουν στην Αταλάντη και θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα δυνατότητα που τους δίνεται, κατά την άποψή σας είναι μεγάλη ή πρόκειται για κάτι το σχετικά περιθωριακό. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους τώρα. Το κύριο Παλέσκης πρώτα απ' όλα, ο οποίος θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε στρατηγέ μου, για αυτή την πάρα πολύ ανοιχτή και ειλικρινή παρέμβαση που κάνατε. Καλό να σας ακούσουμε, διότι κατανοούμε τώρα πολύ καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και πώς η Στρατιωτική Επιτροπή προσπαθεί να λύσει όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η αξιολόγησή σας. Υπάρχουν ακόμη διαφορές μεταξύ των νέων και παλιών κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά τα στρατιωτικά θέματα, την ετοιμότητα για συνεργαστία, την οτροπία που επικρατεί αυτά τα θέματα. Δεύτερη ερώτηση. Οι κλιματικές αλλαγές που μπορούν να προκαλέσουν κάποιες σειράξεις καθώς και τα οικονομικά προβλήματα, η οικονομική κρίση, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε στρατηγέ. Ε, ευχαριστώ στρατηγέ μου, με συγχωρείτε. Ε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το Single European Sky και της Ευρωπαϊκής αεροπορία, Πολεμικής Αεροφορίας από αυτού. Ε, ξεκινήσαμε με την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία απασχόλησε και την ΣΕΝΤΕ μέσω μίας γνωμοδότησης ε, ελέγχθη ότι χρειάζεται ε, καλύτερη προετοιμασία για να μπορέσει να ανταποκριθεί η ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία, πολεμική αεροπορία εις, ε, την, ε, στο επίπεδο τεχνολογίας που υπάρχει. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ένας military deployment coordinator ο οποίος ε, θα μπορέσει να συμβάλλει στην εποπτεία του συστήματος. Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή της πολεμικής αεροπορίας της Ευρώπης στο Single European Sky να διευκολυνθεί με κάποια κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι είχαμε πει στη γνωμοδότηση της ε, υποεπιτροπής μας ότι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό πράγμα το οποίο απέρριψε η Επιτροπή Μεταφορών. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να ε, προετοιμάσουμε σωστά την πολεμική μας αεροπολία και θέτω το ερώτημα ε, ένα τρίμηνο μετά από την ε, αρχή της λειτουργίας του σχετικού κέντρου ε, δηλαδή έχοντας φαντάζομαι ένα είδος μονίμου επιτελείου η κυρία Λέζινγκ Δεν ξέρω αν η ερώτησή μου, η πρώτη μου ερώτηση μπορεί να έχει κάποια απάντηση, αλλά θα πρότεινα να το ε, ε, οριοθετήσουμε πιο σαφώς στο μέλλον διότι μιλήσατε για μία μείωση της ε, στρατιωτικής σημασίας του GSVP ε, και ιδίω σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Θα ήθελα λοιπόν, θα με ενδιέφερε να μου πείτε ε, αν πρόκειται για μία τάξη μεγέθους ή εάν η άποψη αυτή μπορεί να στηριχθεί και με αριθμούς. Θα με ενδιέφερε πολύ. Και επίσης, εάν είναι μία απόφαση των κυβερνήσεων των κρατών μελών που λαμβάνεται σε, ε, στα παρασκήνια. Θα ήθελα να έχω μία απάντηση από αυτού. Επίσης, ο κύριος Ντονζό αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Αταλάντα και θα με ενδιέφερε επίσης πάρα πολύ ε, ποια είναι η προοπτική των δυνάμεων ε, εδάφους ε, στα πλαίσια αυτά και όσον αφορά την αξιολόγηση θα παρακαλούσα να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Ντονζόν δηλαδή σχετικά με τις θέσεις των πειρατών εάν μειώθηκαν κατόπιν της δράσεως της αποστολής Αταλάντα και αν μειώθηκαν σε ποιο χώρο και μπορεί κανείς να καταρτήσει έναν ευρύτερο χώρο όπου δεν έχει υπάρξει μείωση των πειρατικών δραστηριότητων. Δηλαδή επεκτάθηκαν οι επεμβάσεις των πειρατών από τις ακτές σε πιο ευρύ θαλάσσιο χώρο. Υπάρχει μια αξιολόγηση. Θα σας παρακαλούσα να ξεκαθαρίσετε σε ποιο χώρο αναφέρεστε και επίσης αυτός ο ευρύτερος χώρος εάν μπορεί να συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση την οποία θα μας παρουσιάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ μου, έχετε μια πρώτη σειρά ερωτήσεων για να αρχίσει η συζήτηση και μετά θα δούμε αν θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα αρχίσω την πρώτη και τελευταία ερώτηση που αφορά την επιχείρηση Αταλάντη. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε σε πιο ευρύ πλαίσιο. Την προσέγγιση μας προς την ε, ε, πολιτική που θέλουμε να ασκήσουμε στο κέρδος Αφρικής, στη Σομαλία στα πλαίσια του Νέστορ με προσπάθειες αστυνομίας και της ακτοφυλακής και όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην περιοχή με την Κίνα, τον Τζιμπουτί, την Ιεμένη, την ε, Τανζανία. Πρόκειται λοιπόν για ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, λαμβάνουν χώρα όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Έτσι άρχισε και η Αταλάντη και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Πώς θα κάνουν το σχεδιασμό για τις ναυτικές δυνάμεις που έχουν αναπτύξει. Για ένα χρόνο, για πέντε χρόνια. Θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το ξέρουν τα κρατη Αυτό είναι πολιτικά πολύ σημαντικό και για την ε, και επαγγελματική άποψη επίσης. Ποια είναι τώρα η δική μου προσωπική άποψη. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίσουν για το ναυτικό που θα διαθέσει, τις ναυτικές δυνάμεις που διαθέτουν και τα κράτη-μέλη τι θα κάνουν. Τις μεθόδους μας συνεχίζουμε να τις αναπτύσσουμε, να τις ε, αναπτύσσουμε. Ε, έχουμε κάποιες ποιες ε, δυνάμεις ναυτικές τις οποίες έχουμε αποσπάσει σε κάποια εμπορικά πλοία, όχι σε όλα όμως. Αυτό νομίζω όμως είναι πολύ αποτελεσματικό για να καταπολεμήσουμε τους πειρατές και γίνονται και πολύ σημαντικές ε, συζητήσεις με τους ίδιους εφοπλιστές για να έχουμε τις καλύτερες ε, δυνατές επιχειρησιακές ε, πολιτικές που θα εφαρμόσουν για να προστατεύονται τα πλοία μας. Και όσο πληρώνονται So that is problem, but we are dealing with all these things. So it's not just... Λίτρα της τάξης των 100.000 ευρώ κάθε χρόνο δεν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό αφορά του αριθμού νομίζω 10 ή 11 πλοία βρίσκονται στα χέρια των πειρατών 209 πειρα... Ε, ομήρους είχαμε μέχρι χθε και τους τελευταίους 8 μήνες μειώθηκαν σε ποσοστό 40-50%. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους αριθμούς. Η τάση όμως που διαγράφεται τώρα είναι ότι προχωρούμε προς σωστή κατεύθυνση. Και βεβαίως ξέρουμε ότι επεκτείνονται οι επιχειρήσεις μας στην περιοχή αυτή συνέχεια και ακολουθούνται όλο και πιο ακριβείς μέθοδοι. Επίσης, οι περισσότερες επιθέσεις πειρατών γίνονται στον ε, ε, Ινδικό ωκεανό, εκτός του κόλπου και βεβαίως όλα αυτά επηρεάζονται και από τις ε, εποχή των μουσώνων. Τώρα όσον αφορά τις επίγειότητες, στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό για τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα. Και όπως ξέρετε υπάρχει εδώ και δύο μήνες περίπου η απόφαση να αναπτύξουμε και εκεί κάποιες δυνάμεις και θα σας πω ποια είναι η εμπειρία μου. Καταρχάς 15-16 χώρες δέχτηκαν και όσο περισσότερο συζητούσαμε τόσο περισσότερο καταλήγαμε σε συμβιβασμό, σε συμβαστικές λύσεις. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ως εξής τα πράγματα. Στη Σομαλία συνέβαιναν διαφορετικά γεγονότα. Έκλεισε το αεροδρόμιο στο Μογκαντήσιο και με τους υπεύθυνου, με τους επικεφαλείς ε, των στρατιωτικών, των πολιτικών δυνάμεων, της περιφερειακής κυβέρνησης. Συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα είδαμε ποιο θα πρέπει να κάνει τι, ποιο θα πρέπει να προχωρήσει με ποιο τρόπο και είδαν οι συνάδελφοι όταν τους εξηγήσαμε ότι δεν θέλουμε να τους ε, επιβάλλουμε τίποτε, Απλώ θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έτσι ήταν η αντίδρασή τους, τους ε, πολύ θετική. Μιλήσαμε για τον κίνδυνο παράπλευρων ε, ζημιών και τελικά το σχέδιο που προτείνουμε έγινε αποδεκτό και τώρα έχουμε θέση, θέσαμε πριν από έξι εβδομάδες ε, σε εκκίνηση το πρώτο πρόγραμμα αντεπίθεση θα θέλετε και πρέπει να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ επιτυχείς. Τώρα, με μεγάλη προσοχή κάνουμε αξιολόγηση αυτής της επιχείρησης. Υπάρχει ενδεχομένως κίνδυνος να τραυματίσουν κάποιους ομήρους οι ε, πειρατές που είναι και πολύ έξυπνοι, ευφυείς και βρίσκουν νέες μεθόδους και προσαρμόζονται σε αυτά τα οποία κάνουμε εμείς. Αλλά πρέπει να πω ότι μετά από την πρώτη μας πηδήση μαθαίνουμε από αυτά τα οποία έγιναν και προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια νέα πολιτική. Αυτό αφορά την Αταλάντη. Τώρα, το θέμα που αφορά την ε, κατάσταση την οποία έχουμε μετά τη τελευταία διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγική της Ευρώπης του 2003 ήταν πάρα πολύ, ε, έδωσε πάρα πολύ καλές ε, οδηγίες και τρόπο με τον οποίο έπρεπε να ενεργήσουμε για την πρόληψη σειράξεων, για τον ανθρωπιστικό ε, τομέα, για να μπορέσουμε να κάνουμε επιχειρήσεις εκενώσεων, διάσωσης κτλ. Επίσης, Πρέπει να πω ότι οι ομάδες που διαθέτουμε βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν προβλήματα με τον προϋπολογισμό και έτσι η ετοιμότητα κατά κάποιο τρόπο αμβλύνεται δεδομένου ότι κοστίζει. Είναι δαπανηρή. Μεταξύ των κρατών μελών βλέπω να υπάρχει θετική άποψη για αυτό το θέμα. Ένας τρόπος είναι το pooling and sharing για να μπορέσουμε μέσα και δυνατότητες να τα μοιραστούμε. Υπάρχει όμως και ένα αντιφατικό στοιχείο. Όσο περισσότερη πίεση ασκείται σε μεμονωμένα κράτη-μέλη, αντί να υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και να πει κάποιος αντί να έχω τίποτα, ας έχω κάτι, η τάση είναι να γίνεται κανείς πώς, ε, περισσότερο εσωστρεφής για να επιλύσει το πρόβλημά του. Και αυτό δεν είναι κάτι το θετικό. Υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση. Και πιστεύω ότι πραγματικά με την κατάλληλε ηγετικέ μορφέ μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ, το συζητούμε το πρόβλημα. Για μας το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει και ο Βόρειος Πόλος και η Αρκτική και η Ευρώπη. Ξέρουμε ότι οι λαγέ κλιματικές θα αλλάξει και σημαντικά τον τρόπο τον οποίο ενεργούμε και στις διάφορες υπήρους. Και είμαστε σε μία πρώτη φάση. Δεν υπάρχει μυστικό πλέον το ότι αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι ε, στην βορειότερη ε, ε, μέρος της Ρωσίας αναπτύσσουν κάποιες δυνάμεις και εμείς παρακολουθούμε με προσοχή το τι ακριβώς κάνουν. Κάτι άλλο που έχει σχέση με τις κλιματικές αλλαγές είναι το ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τις ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας και άμβληση των προβλημάτων σε περίπτωση καταστροφών κλιματικές αλλαγές είναι λοιπόν πολύ σημαντικές. Και εδώ και ξέρουμε ότι πολλές φορές δημιουργήθηκαν ε, δυσκολίες μεταξύ του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους της βοήθειας. Νομίζω όμως ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρωπιστικό πρόβλημα και κυρίως για να προστατεύσουμε και τα χρήματα των φορολογουμένων δεν φιδόμεθα προσπαθειών. Όσον αφορά τον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ίσως πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα και σημαντικά προγράμματα τα οποία συνεχίζονται και θα συνεχιστούν να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια. Στην ε, Στρατιωτική Επιτροπή είχαμε από κοινού συζητήσεις με την Επιτροπή και συναντήσεις μάλλον με την Επιτροπή. Δύο φορές θέσαμε το θέμα σε όλους τους επικεφαλείς των Υπουργείων Άμυνας για το θέμα αυτό, ώστε να έχουμε την εγγύηση ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα σχέδια για τον ενιαίο ευρωπαϊκό Κορονό όλες οι διαστάσεις των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, η κατάρτιση και η ελευθερία χρησιμοποίησης του ευρωπαϊκού νιέ ουρανού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και με απογοήτευσε την τελευταία στην τελευταία συνέντευξη όταν θέσαμε το θέμα το ότι όταν συζητάτε το θέμα αυτό, τουλάχιστον μόνο καμιά δεκαετία χώρες είναι παρούσες. Πρέπει λοιπόν να σπρώξουμε τα πράγματα ώστε όλοι οι επικεφαλείς να συνειδητοποιήσουν περί ως πρόκειται. Η συνεργασία στην τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει όλοι οι μετέχοντες να καταλάβουν ότι δεν έχει μόνο κόστος αυτό το εγχείρημα, αλλά έχει και μεγάλα ωφέλη. Βραχυπρόθεσμα υπάρχει κόστος, αλλά μέσο και μακροπρόθεσμα θα βοηθηθούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά το Center, το επιχειρησιακό κέντρο, το έθεσε το θέμα και το πρόεδρος. Έγιναν εκτενέστατες πολιτικές συζητήσεις. Μιλούμε για πάρα πολύ λίγα άτομα, 12 προς το παρόν. Βρήκαμε τρόπο αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει μετά από έξι μήνες και προσωπικά πιστεύω ότι ο στόχος είναι δηλαδή να υποστηρίξει και να συντονίσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο κέρας της Αφρικής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, θα πω ότι σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για πολιτικό θέμα. Γι' αυτό δεν θα πω τις απόψεις μου, θα πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε τι έχει γίνει τους τελευταίους μήνες σε σχέση με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έτσι κάλυψε τις περισσότερες ερωτήσεις. Ίσως έχω μία αυτό το αυτό που είπατε ότι είναι κάποια ερώτηση στην οποία δεν βλέπουμε δυνατή λύση. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Υπάρχουν όμως μεγάλες δυσκολίες. Μιλήσατε στα πλαίσια της ΚΕΠΑ για το ρόλο του ΝΑΤΟ. Η ισχύ της Ευρώπης στον τομέα αυτό είναι ότι μπορούμε να είμαστε ε, πάρα πολύ ενεργοί σε όλα τα στάδια, ακόμη και σε αρχικό στάδιο, για να μπορέσουμε να προλάβουμε μία σύραξη. Έχουμε τα μέσα. Το 2006 στην Κινσάσα, με τις εκλογές κάναμε κάτι τέτοιο, είχαμε ε, μέσα για να ενεργήσουμε το στρατιωτικό η στρατηγική διάσταση ήταν επίσης παρούσα. Θα υπενθυμίσω επίσης το παράδειγμα του Κονγκό όπου είχαμε παρουσία με ειδικέ δυνάμεις και είμαι σίγουρος ότι έτσι αποφύγαμε τη γενοκτονία. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να μπορέσουμε να κάνουμε πρόληψη των σειράξεων σε αρχικό στάδιο. Διότι εάν δεν ενεργήσουμε έγκαιρα και ξεσπάσει η σύραξη, είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Το ΝΑΤΟ βεβαίως ένα άλλο στάδιο μπορεί να διαθέσει τα μέσα που. Εμείς όμως κάνουμε, ενεργούμε διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει διαχωρισμός του τρόπου δράση και ενέργειας. Αλλά πρέπει να πω ότι και το ΝΑΤΟ έχει πολύ καλές δυνατότητες. Και όταν φτάσει στο ανώτατο όριο η σύραξη και μετά πέσουν οι εντάσεις και πρέπει να γίνει ε, η ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση της ε, κοινωνίας και όλων των προσπαθειών που πρέπει να καταβάλουμε για να ξανασυσταθεί μια κοινωνία σε όλους τους τομείς, εκεί είμαστε. λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με σύραξη μπορούμε να κάνουμε καταμερισμό των ε, ε, δράσεών μας ο καθένας. Και βεβαίως εκεί είμαστε για να ανακουφίσουμε τον πληθυσμό, για να κάνουμε διάφορες επιχειρήσεις, διάσωσης και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε στρατηγή κυρία Λέζινγκ. Θέλατε να πείτε κάτι. Έχω δύο ακόμη ερωτήσεις για διευκρινήσεις. Καταρχήν όσον αφορά την αξιολόγηση της αποστολής Αταλάντα μιλήσατε για τη διεύρυνση του πεδίου των επιχειρήσεων και για μία μείωση κατά 40 έως 50%. Συγκεκριμένη ερώτηση. Η μείωση 40 έως 50% αναφέρεται σε αυτό το διευρυμένο χώρο επιχειρήσεων ή σχετικά με αρχικό, με το αρχικό πεδίο επιχειρήσεων. Αυτή τη διευκρίνηση θα ήθελα παρακαλώ και μετά όσον αφορά τις ε, δυνάμεις ξηράς. Είπατε ότι ε, μπόρεσε κανείς να καταστρέψει τα πλοία των πειρατών. Εγώ δεν είμαι ειδική όμως, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ότι πρόκειται ε, για πλοία των πειρατών και όχι για ψαράδικα ή πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια τέτοια επέμβαση. Πριν απαντήσω, ο κύριος Μπαλτιέρη ήθελε να σχολιάσει και να ρωτήσει κάτι. Ευχαριστώ, στρατηγέ. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση σας άκουσα εδώ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε πάλι μαζί μας. Ήθελα απλά να μοιραστώ μια αίσθηση που μου δημιουργείται πολιτικής γενικής φύσης όταν σας ακούω σκεπτόμενος τα όσα έχει πει αυτό το κοινοβούλιο και γράψε πέρυσι, τους περασμένους μήνες και με βάση του στενού διαλόγου με εσάς και με τη Στρατιωτική Επιτροπή και δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης. Αντιλήφθηκα από τα όσα μας λέτε έναν ε, τον, δεν θα έλεγα απεσιόδοξο ακριβώς, ε, απογοητευμένο, αλλά κάπως ρεαλιστικό όσον αφορά την αξιολόγηση του γεγονότος ότι κατά πόσο αυτές οι δυνατότητες που έχουμε προσδιορίσει τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο πλαίσιο των παγκόσμιων εξελίξεων, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η κρίση και κατά πόσο όλα αυτά επιβάλλουν ένα ρόλο πολύ ισχυρό. Μου φαίνεται ωστόσο ότι πολιτικά τα αποτελέσματα σε όλα τα μέτωπα που αναφέρατε κι εσείς ε, ο στρατηγικούς κοινούς ε, στόχους, οικοδόμηση ικανοτήτων, κοινών, και μεγαλύτερο συντονισμό τη διαδικασία σχεδιασμού σε όλε αυτέ τι πτυχέ. Εν τέλει, υπάρχει ένα κενό μεταξύ των δυνατοτήτων και των πολιτικών δεσμεύσεων εκ μέρου των κρατών μελών που θέτουν κάποια βαθιά ερωτήματα σε όσου ε, πιστεύουν στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ε, η ερώτησή μου δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή ή ε, συγκεκριμένη, αλλά θα θεωρώ ότι μια οποιαδήποτε αξιολόγηση αυτή τη στιγμή θα είναι ιδιαίτερα επικριτική και προβληματική. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη ηγεσία, περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερες προτάσεις, περισσότερο θάρρος. Μου φαίνεται ότι οι δυσκολίες που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κρίσης αποτυπώνονται και σε αυτό το μέτωπο. Αναρωτιέμαι λοιπόν με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε ξανά αυτόν τον ενάρετο κύκλο μεταξύ των στρατηγικών στόχων πέραν της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας με κοινή χρήση δυνατοτήτων και διαδικασιών ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ σας αφήνω το λόγο για τα τελευταία σας λόγια ε, να απαντήσετε στην κυρία Λέζιν και στον κύριο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την αξιολόγηση του Αταλάντα, οι αριθμοί δεν σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με την επέκταση της περιοχής ε, δράσης. ευχαριστώ θα σας δώσω ακριβώς τα μεγέθη για το ποια ήταν η εξέλιξη, η ανάπτυξη της τελευταίους 8 μήνες. Μπορώ να το πράξω αμέσως. Το δεύτερο κομμάτι του ερωτηματός σας σε σχέση με την αντιμετώπιση των πειρατών και πώς γνωρίζουμε ότι στοχεύουμε τα σωστό στόχο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε ιδιαίτερα ακριβείς πληροφορίες και εικόνες, φωτογραφίες με πολλές λεπτομέρειες και έχουμε προσέξει ιδιαίτερα την ελαχιστοποίηση οποιοδήποτε παράπλευρου κινδύνου ζημίας. Τα προβλήματα logistics είναι πολύ απομακρυσμένα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς λειτουργούν. Προσπαθούμε να πλήξουμε το υλικό τους, την υποδομή τους και όχι ανθρώπους. Η ανάλυση των εικόνων που έχουμε μας βοηθάει να ακολουθούμε διαδικασίες επιμέρους μεμονωμένες σε αυτού του ίδιου στις δραστηριότητες δεν υπάρχουν διασφαλίσεις ούτε εγγύησει. Αλλά για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε εστιαστεί ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη προσοχή και προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε. Η δεύτερη ερώτηση το πώς βλέπουμε το μήνυμα του Κοινοβουλίου το συζητάμε συνεργαζόμαστε με το PSC, έχουμε μόνιμη έδρα στο PSC για να είμαι πιο συγκεκριμένο η μελέτη του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις δημοσιονομικές περικοπές την υποστηρίξαμε, συμβάλαμε σε αυτήν και μας ήταν και εξαιρετικά χρήσιμη. το ζήτημα των στρατηγικών στόχων, των ικανοτήτων και του συντονισμού και του σχεδιασμού. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα κλειδιά. Ταξιδεύοντας στα διάφορα κράτη-μέλη, οι 27 αυτές χώρες λαμβάνουν 27 μεμονωμένες επιμέρους αποφάσεις για κάθε περίπτωση και όταν κάποια κράτη-μέλη λαμβάνουν τις ίδιες αποφάσεις για συγκεκριμένες ικανότητε ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς κανένα συντονισμό και χωρίς καμία ικανότητα. Αυτός ο συντονισμός λοιπόν μεταξύ των 27 διαφορετικών αποφάσεων είναι κάτι που πρέπει να αρχίσει να γίνεται. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Να σας επαναλάβω ότι αυτό το ζήτημα τώρα αφορά τους επικεφαλείς, ε, του αρχηγούς κρατών και χαίρομαι που θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα του Συμβουλίου για το επόμενο έτος. Αυτή η ατζέντα θα πρέπει να συζητηθεί. Καταλαβαίνω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά αυτό το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας των επιμέρους κρατών μελών ε, όταν ε, προβαίνουμε σε pooling and sharing υψηλού επίπεδου είναι και θέμα αμυντικής βιομηχανίας πώς μπορούμε να συντονίσουμε την αμυντική βιομηχανία και επίσης υπό το ίδιο πνεύμα και απασχόληση και η εφαρμογή όλων αυτών. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, είναι ζήτημα μαθηματικών. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Έχουμε την πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε σε συνταρακτικές αλλαγές ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ίδιες διαδικασίες με, όπως αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ στρέτηγε για τις διευκρινήσεις σας. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Μας δίνουν πολλές πληροφορίες και για τις δικές μας ε, συζητήσεις. Εσείς εγκαταλείπετε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να έχουμε και μια τελευταία ανταλλαγή απόψεων είτε τη στιγμή της αναχωρησής σας ή ενδεχομένως μετά αφού θα διατηρείτε την εμπειρογνωμοσύνη και ένα μάτι ε, εμπεριστατωμένο σε θέματα πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες. Ε, είναι βέβαιο ότι ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτεται σήμερα θα πρέπει να οδηγήσουν σε κάποιες αποφάσεις πιο σημαντικές από αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα, ειδικότερα από τα κράτη-μέλη αλλά και από, τη, από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλήθεια είναι ότι η τελική απόφαση σε θέματα άμυνας αναποκτέω ουσιαστικά αποκλειστικά στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο, αλλά διαπιστώνουμε ωστόσο συνέβη στην περίπτωση της Λιβύης και το αναφέρετε και εσείς από το 2008 καμία στρατιωτική, πραγματική στρατιωτική επιχείρηση εκτός από τη UTM Σομαλίας δεν ξεκίνησε βλέπουμε ότι οι δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ίδιες αυτές τις δομές, ορισμένες φορές διστάζουν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για μια τεράστια ευθύνη τόσο για τα κράτη-μέλη όσο και για τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ειδικότερα σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε να λάβουμε αυτές τις αποφάσεις που θα είναι απαραίτητες και ούτως ή άλλως ε, η δημοσιονομική κρίση θα μας, ε, θα μας το επιβάλλει ανεξάρτητα από τη βούληση των κρατών μελών. να δούμε λοιπόν αν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη μια συνάντηση μαζί σας το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σα Σας προτείνω ε, για 10 λεπτά, το πολύ πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, το GMS, e να επανέλθουμε και να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο θέμα το οποίο είχε προεδρεύσει ο κ. Μαυρονικόλας και το οποίο αφορούσε το Horizon 2020. Ακούσαμε κάποια σχόλια, κάποιες ερωτήσεις από συναδέλφους. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ε, θα μπορούσε να απαντήσει στα σχόλια που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Ο κ. Σαλακάν από την ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις στα γρήγορα. Θα ήθελα να επαναλάβω την πρόταση της Κομισιόν για τα θέματα ασφαλείας. Αναφέρεται πράγματι αρκετά ρητά για πρώτη φορά στην κοινή πολιτική, στην κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Ταυτόχρονα παραμένει μια ρητή αναφόρα για ολόκληρο το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο του ορίζοντα 2020 όσον αφορά την αποκλειστικά μη στρατιωτική πτυχή ε, του προγράμματος πλαισίου και της έρευνας, της μη στρατιωτικής έρευνας. Αυτές οι δύο δεν έρχονται σε αντίφαση κατά την άποψή μας. Ουσιαστικά η ίδια προσέγγιση αποκλειστικά μη στρατιωτική υπάρχει ήδη στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και αυτό δεν μας εμπόδισε να ξεκινήσουμε και να ενισχύσουμε μια πολύτιμη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας σε διάφορους τομείς όπως η ασφάλεια από τυχόν χημικές, βιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις από τη χρήση ε, εναρίων μέσων ε, μη επανδρομένων, η θαλάσσια επιτήρηση, οι θεμελιώδεις τεχνολογίες για ανεξαρτησία ατομής, στους οποίους εργαζόμαστε εδώ και χρόνια με τους συναδέλφους ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας καθώς και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τις οικονομικές πτυχές των διαφόρων μορφών έρευνας όπως υπόθηκε από διάφορους ε, Ε, ήδη βουλευτές ε, προηγουμένως ε, η έρευνα στον τομέα της άμυνας είναι πολύ ανώτερη από όσο μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα πλαίσιο. Από άποψη λοιπόν προσθέμενης αξίας συμφωνούμε όσον αφορά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να εντοπίσουμε σημαντική προστιθέμενη αξία σε έναν τομέα όπως την στρατιωτική αμυντική έρευνα. Αντιθέτως, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, σήμερα ο υπολογισμός στα κονδύλια που δαπανώνται στο πρόγραμμα πλαίσιο ισούνται χονδρικά με το 50% το μισό δηλαδή του ό,τι δαπανάτε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για την έρευνα σε πολιτικά θέματα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όχι μόνο είναι σημαντική η προστιθέμενη αξία, αλλά και ότι η έρευνα ε, είναι ιδιαίτερα επικοδομητική για τον μη στρατιωτικό τομέα. Αποτελεί επικοδομητική συνιστόσα. Ήθελα επίσης να αναφέρω αυτό το οποίο εμάς πρακτικά απόψη υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος πλαισίου και σε θέματα ασφαλείας. Αυτό που εμάς μας φαίνεται ότι είναι ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μιλάμε για το πρόβλημα συνεργασίας, απευθείας συμμετοχής του πλευράς της τη ευρωπαϊκή αγορά πολιτική προστασία, η βιομηχανία, ο τομέας παραγωγή νέων τεχνολογιών έχει ήδη διεξάγει αρκετές εργασίες προσαρμογής και βελτιστοποίησης. Ενώ από την πλευρά της ζήτησης η αγορά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά κατακαιρματισμένη σε ουσιαστικά 27 εθνικές αγορές. Συχνά παρατηρείται επίσης δυσκολία εκ μέρους των εθνικών αρχών να αξιολογήσουν επαρκώς ε, τη σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο όπου η κοινωνία των πολιτών ε, αναρωτιέται όλο και περισσότερο κατά πόσο είναι εφαρμόσιμες ορισμένες τεχνολογίες, τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι τεχνολογίες στην ζωή των πολιτών, στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ιδιωτική του ζωή. Κατά την άποψή μα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια δημοκρατική συζήτηση για την εφαρμοσιμότητα αυτών των τεχνολογιών και για τη δυνατότητα και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από μια ενδεχομένως μια μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών αρχών σε αυτή την τεχνολογική προσπάθεια. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει τη στενή και εντατική συνεργασία και με τις εθνικές αρχές ε, σε θέματα άμυνας. Θεωρούμε ότι ήδη στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, όπως και στον επόμενο ορίζοντα 2020, η υλοποίηση ενός προγράμματος έρευνας μπορεί να διευκολύνει αυτές τις συναντήσεις, αυτούς τους συντονισμούς, αυτή τη δημοκρατική συζήτηση στην οποία αναφέρθηκαν οι, οι συναδελφοί σας προηγουμένως. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρέον από την υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζοντας, θα ήθελα να Βεβαίως αυτά τα οποία είπε για την συνεργασία ο συναδελφός μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας επέτρεψε να έχουν πάρα πολύ καλό συντονισμό στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΦΣΕ, τον τομέα της άμυνας. Δόθηκαν κάποια παραδείγματα καρποφόρου συνεργασίας και αυτό το οποίο έχουμε θέσει σε, σε κίνηση τώρα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι κάτι το οποίο είναι και στα, γίνεται και στα πλαίσια του ορίζοντος 20 σε, σε Σήμερα το πρωί αναφέρθηκε η κυβερνοασφάλεια, ε, που είναι ένα εγκάρσιο θέμα και αφορά τους πάντες. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή καταρτίζουν στο θέμα αυτό κοινή πολιτική και στο θέμα του διαστήματος και θα συζητηθεί σε λίγο το θέμα αυτό. Σε αυτούς τους τομείς έχουμε τις key enabling technologies, τεχνολογίες εχμής κλειδιά που μας επιτρέπουν να βρούμε κοινέ εφαρμογές για στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ε, εφαρμογές. Αυτά είναι λοιπόν θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την άμυνα αλλά και το διάστημα. Και συνεργαζόμαστε το τομέα αυτό και με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Είναι όλα αυτά θέματα στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρχει κοινή προσέγγιση μεταξύ της Επιτροπής και των Υπουργείων Άμυνας. Αυτό προσδίδει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και δεν πρέπει να παραγνωριστεί ως χαρακτηριστικό. Για όλους αυτούς τους λόγους υποστηρίζουμε πλήρως την έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, ώστε να παγιωθεί και να διαρθωρθεί καλύτερα αυτή η κοινή προσέγγιση ώστε να έχουμε κοινά ωφέλη στους δύο αυτούς τομείς που μας απασχολούν από κοινού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο τελευταίες παρεμβάσεις για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, κυρία Λέζιν και κύριος Γκάλλον. κυρία Λέζιν πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλια του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται πολύ ενδιαφέροντα και γελάω διότι είπε ναι μεν ε, υπάρχει έρευνα η οποία απευθύνεται στον πολιτικό χώρο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά χρησιμοποιήθηκε στον πολιτικό χώρο. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να ξέρουμε ακριβώς ε, σε τι απευθύνεται η έρευνα και όχι ότι θα υπάρχουν και πολιτικές ε, επιπτώσεις και εφαρμογές απλούστατα να ξέρουν συγκεκριμένα οι πολίτες και να υπάρχει διαφάνεια για το τι είναι η χρήση η οποία γίνεται. Ο κύριος Γκάλερ, μόνο μία φράση. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σαφήνειά του, διότι νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω πλήρως όπως και με τον εισηγητή. Νομίζω ότι έχουμε μία καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία. Ευχαριστώ. Κύριε Μαυρονικόλα, θέλετε εσείς να εμπλουτίσετε τη συζήτηση και να την κλείσετε τώρα. Αυτό που είπα προηγουμένως. Υπάρχουν ορισμένες ε, αντιρρήσεις στην έκθεση. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε μία γλωσσική προσέγγιση η οποία θα διασκεδάσει ορισμένες από αυτές τις αντιρρήσεις, πράγμα που μπορεί να γίνει ίσως με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου αρχές Σεπτεμβρίου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο έθεσαν το πρόβλημα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε. Δεν θυμάμαι πλέον τις επόμενες ημερομηνίες, ε, τις προθεσμίες για αυτή τη γνωμοδότηση. 23 Αυγούστου προθεσμία για υποβολή τροπολογιών για μια νέα συζήτηση στα μέσα του μήνου Σεπτεμβρίου στην ΣΕΝΤΕ. Περνάμε στο επόμενο θέμα με τους ίδιους ομιλητές ε, ένα θέμα σημαντικό που αφορά το σύστημα GMS αυτό το σύστημα γεωσκόπησης, παρατηρήσει της γης που έχει φυσικά εφαρμογές σε θέματα ασφαλείας και άμυνας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στη στρατηγική στρατηγική λήψη αποφάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και τον Γαλιλαίο ένα πρόγραμμα το οποίο ωστόσο βρίσκεται υπό απειλή αυτή τη στιγμή από άψη χρηματοδότησης Οι θέσεις για αυτό το πρόγραμμα διαφέρουν ε, στο Κοινοβούλιο. Έχει υπενθυμιστεί σε πολλά ψηφίσματα με τελευταία ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου του 2012 ότι η προσήλωσή του σε μια κοινοτική χρηματοδότηση αυτού του μέσου στην ανακοίνωση της Κομισιόν ε, και στη συζήτηση του Συμβούλιο βλέπουμε άλλες εναλλακτικές που δεν είναι ιδιαίτερα δεν αντιμετωπίζονται ευνοϊκά από το Κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφωνία και θα θέλαμε τώρα να σας παρουσιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση με την Κομισιόν ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε. Ο κύριος ε, Αλακαρνέ, έχετε το λόγο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, την Επιτροπή για αυτή τη συζήτηση και να υπενθυμίσω την τρέχουσα θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το GMES. Δεν περιλαμβάνει το GMS e τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό καταδείχθηκε σαφώς στην πρόταση της Κομισιόν για τον νέο προπολογισμό που έγινε τον Ιούνιο πέρυσι. Μέσα σε αυτή την, πρώτη, αυτή την πρόταση ακολούθησαν δύο ανακοινώσει συγκεκριμένα για το ζήτημα του GMS. Σε αυτές τις ανακοινώσει η Κομισιόν απευθύνθηκε κυρίως στα κράτη-μέλη ώστε να του ζητήσει να λάβουν σαφή θέση όσον αφορά μια δικυβερνητική προσέγγιση για το GMS. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι μια συζήτηση εντός του Συμβουλίου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και άλλων συμβουλίων γενικών υποθέσεων είναι αρκετά ζωηρές οι συζητήσεις. Πρόσφατα η Προεδρία, η προηγούμενη Προεδρία της Δανίας είχε θέσει το GMS σε ένα negotiating box, σε ένα κουτί διαπραγματεύσεων με μία μόνο επιλογή, την επιλογή της επανένταξης του GMS εντός των δημοσιονομικών προοπτικών. Εμείς υπομονούμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή υπό την τρέχουσα Κυπριακή Προεδρία και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σημειώσει τις όποιες πιθανές θέσεις και τις όποιες ανακοινώσεις, οι επίσημες δηλώσεις του Συμβουλίου, ειδικότερα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Bien, Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκολτιέρη μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δυσκολία μπορώ να καταλάβω τη λογική που στηρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή μάλλον μπορεί να την καταλάβει κανείς με τη μέγιστη καλή θέληση. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μια βούληση προστασίας ενός τόσο σημαντικού μέσου από τους κινδύνους ε, μιας δημοσιονομικής διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, το, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην καλύτερη των υποθέσεων, το αποτέλεσμα μιας τέτοιας βούλησης ε, υπεράσπισης, προστασίας ενός τόσο θεμελιώδους προγράμματος ε, όπως το GMES ενέχει τον κίνδυνο κατά την κρίση μου αφενός να επιτείνει τους κινδύνους αφετέρου να οδηγήσει σε μια αντίφαση αδύνατη σε αυτό το κοινοβούλιο διότι πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο Πρέπει να γίνει αυτό γιατί πρέπει να βγάζουμε κομμάτια από τον προπολογισμό ώστε να τα ξαναβάζουμε μετά. Αυτό είναι παράδοξο. Εάν θεωρούμε ότι η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει τις τρέχουσες κρίσεις συνεχίζοντας να οικοδομεί μορφές outsourcing του ίδιου της του εαυτού ακόμη και όταν Δεν υπάρχουν λόγοι, δεν έχουμε βέτο, δεν υπάρχουν εξαναγκασμοί κρατών μελών. Υπάρχει το δημοσιονομικό σύμφωνο για παράδειγμα, υπάρχει κάποια λογική, αλλά εδώ πάμε να παίρνουμε πόρους από κάπου και να τους βάζουμε αλλού. Ουσιαστικά αυτό το κοινοβούλιο φυσικά αντιδρά. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μια πρόκληση. Και έτσι αφαιρείται και οποιαδήποτε εγγύηση για το μέλλον του GMS. Μιλάμε για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης. Μιλάμε για τη δεύτερη φάση ενός πράγματος που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που βγαίνουν από τον προπολογισμό και ξαφνικά ξαναμπαίνουν από το παράθυρο σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για το GMS ε, ε, για την Αφρική κατά ε, είναι μια απαράδεκτη λύση που θα μπορούσε να οδηγήσει να δυσκολέψει, να δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, οδηγώντας έτσι σε κοινοβουλευτικά αντίπεινα κατά κάποιο τρόπο για άλλα ε, assets του προϋπολογισμού και υπονομεύοντας την κοινή ε, προσπάθεια του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για τη διασφάλιση του επαρκούς κατακαιρματισμού των πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τη συγκεκριμένη εδώ επιτροπή από πολιτική και στρατηγική, ε, όσον αφορά την ανάπτυξη αυτή τη ικανότητα, εμεί την υποστηρίζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια υποδομή ευρωπαϊκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πνεύμα υπό το οποίο έχουμε δεσμευτεί και στο παρελθόν στις συζητήσεις μας ε, να ευνοήσουμε τη συμβολή του προπολογισμού και στις πολιτικές ασφαλείας. Ταυτόχρονα ακριβώς γι' αυτό το θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα τέτοιο ε, ουσιαστικό πλεονέκτημα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάλερ. Ευχαριστώ. Βασικά συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος Γουαλκέρη, Δηλαδή είναι ουσιαστικά θέμα αρχής και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να προτείνει ε, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα διαχειρίζονται διακυβερνητικά. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει ορθά. Και αυτό όχι μόνο διότι πλέον θα είναι εκτός ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι θέμα αρχής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά εις το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προτείνεται την Προεδρία έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις θέσεις συμβούλων τα κράτη. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, καμία συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας υπενθυμίζω ότι στις 16 Φεβρουαρίου σε ένα ψήφισμα επί του θέματος είχαμε πει και διαβάζω αγγλικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πιστεύει ότι το ε, οικονομικό GMES μπορεί να λειτουργήσει ε, βιώσιμα ε, σύμφωνα με το πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή το είχαμε δηλώσει ρητός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να ξανασκεφτούν εάν θα συνεχίσουν επ' αυτής της οδού ή όχι. Η κυρία Λόιζινγκ, χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι λόγοι για τους ε, οποίους ε, αφαιρέθηκε από το δημοσιονομικό πλαίσιο διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούσε για την περίοδο 14 μέχρι 2020 για 5,841 δις και αντιλαμβάνομαι ότι ο κόστος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο διότι ε, το, ε, σε μια ε, επιστολή του Γερμανικού Κέντρου Αεροπλοείας λέγεται ότι μπορεί να υπήρχαν τέτοιες τεράστιες δαπάνες που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύω λοιπόν ότι η διάσταση αυτή θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ανοιχτά ε, και να συζητηθεί. Επίσης επανέρχομαι σε ένα παρεμφερές θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, δηλαδή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 ε, πολιτικές και ε, στρατιωτικές χρήσεις όπου λέγεται πως ε, οι διτές δυνατότητες παρακολουθήσεως δηλαδή και πολιτική και στρατιωτική μπορούν να συμβάλλουν σε το χρήση του GMES πράγμα το οποίο δεν προϋποθέτει ότι θα πρέπει υπό αυτές τις προϋποθέσεις να χρηματοδοτηθεί το θέμα από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βέβαια ε, μπορεί να μου λεχθεί ότι ε, αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν και έχουν ε, χρησιμοποιηθεί γραμμές του προπολογισμού και στο παρελθόν στο αυτό το πλαίσιο. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω να επανέλθουμε με μεγάλη διαφάνεια σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο διαπιστώσεις ε, τεχνικές ε, και συγκεκριμένων συμβάντων ήθελα να κάνω. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε για το μέλλον αλλά μέχρι στιγμής το πρόγραμμα GMES δεν αυξάνει τα κόστη του. Σε περίπτωση που προκύψουν δαπάνες προσαρμογής των υποδομών σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τότε μιλάμε για αυξήσεις δαπανών που αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στο 1% ούτε καν. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που λέμε συνήθως για τα μεγάλα έργα υποδομής. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα πώς γίνεται αυτό το πρόγραμμα σημαντικό πρόγραμμα υποδομών να προτείνεται να μην συμπεριληφθεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας επαναλαμβάνω αυτό που λέει η επίσημη ανακοίνωση. Ο ουσιαστικός, ο βασικός λόγος είναι η προσωρινή, η χρονική μάλλον διάσταση τέτοιων προγραμμάτων που δεν συντονίζονται με τον χρηματοδοτικό κύκλο των κοινοτικών δαπανών. Για να τελειώσω, ήθελα επίσης να απαντήσω στην πολύ καλή παρατηρήση της κυρίας Λέζινγκ σε σχέση με την πιθανή χρήση του GMES για στρατιωτικές χρήσεις. Θα ήθελα να σας επισημάνω απλά ότι η διαστημικές κυρίως υποδομές τις οποίες βασίζεται το GMS για να παρέχει τις υπηρεσίες του αναφέρομαι δηλαδή στους δορυφόρους που ονομάζονται Sentinel φρουροί οι, πρώτοι ελπίζουμε, οι πρώτοι ελπίζουμε θα εκτοξευτούν του χρόνου τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά δεν σχετίζονται με στρατιωτικές έρευνες για να σας εξηγήσω η, περι, η βέλτιστη περιφόρα που μπορεί να επιτευχθεί με αυτούς τους δορυφόρους ή μάλλον συγγνώμη η ανάλυση των εικόνων η ανάλυση των εικόνων που μπορεί να επιτευχθεί με αυτούς τους δορυφόρους είναι μέτρων ενώ οι στρατιωτικοί δορυφόροι ε, έχουν ανάλυση μέχρι εκατοστών. Φυσιολογικά λοιπόν όταν μιλάμε για στρατιωτικές εφαρμόγες ε, στους δορυφόρους, μιλάμε για δορυφόρους που χρησιμοποιούν πολύ πιο προηγμένες τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γκουαλτιέρη, θέλω να πάρει το λόγο. ότι η απάντηση που μας δίνεται εντείνει τις αμφιβολίες μας. Ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω από τεχνικής άποψης τι σημαίνει ότι η αιτία για την οποία δεν συμπεριλαμβάνεται είναι ότι οι διαστάσεις του, το μέγεθός του και η διάρκεια του δεν συμβαδίζει με το δημοσιονομικό, με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μιλάμε για επταετής δημοσιονομικές προοπτικές που περιλαμβάνουν πολιτικές με πόρους πολύ υψηλότερους από τους πόρους του GMS. Πολιτικές πιο περιορισμένης χρονικής εμβέλειας και που θεωρείται ότι θα χρειαστούν υποστήριξη και αργότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η, η Επιτροπή, το προσωπικό της, τα κτίρια, όπως και συγκεκριμένες επενδύσεις. Εξάλλου στο σχέδιο της διακυβερνητικής απόφασης λέγεται ότι τα κράτη-μέλη θα καλύπτουν το Ταμείο GMES από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Οθετείται δηλαδή ακριβώς η ίδια περίοδος με αυτή των δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά λέμε ότι ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός δεν συμβαδίζει, διότι είναι επταετής και μετά ε, δίνουμε κάτι για 7 χρόνια. Τα ίδια 7 χρόνια που θα χρηματοδοτήσουν τα κράτη-μέλη με τα ίδια χρήματα που θα μπορούσαν να βάλουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματο. Εγώ πραγματικά λοιπόν δυσκολεύομαι να καταλάβω από τεχνική και πρακτική άποψη τη λογική, τη νόημα αυτού του επιχειρήματο που μόλι μα παρουσιάσατε. Bien, θα θέλατε να απαντήσετε. Όχι, θα μείνουμε σε αυτό. Πολύ καλά. Νομίζω ότι εκφράστηκαν με σαφήνεια οι διάφορες τοποθετήσεις. Οι συνάδελφοι εξέφρασαν ποια ήταν και η θέση του Κοινοβουλίου που στο ψήφισμα του Φεβρουαρίου 2012 επίσης είχε εκφραστεί με σαφήνεια. Περιμένουμε λοιπόν τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ όλους σήμερα το απόγευμα. Στο μενού τι έχουμε. Την κλιματική αλλαγή, την PSDC, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και γνωμοδότηση για τα εξωτερικά σύνορα από την κυρία Φλότρο. Και θα τελειώσουμε με συνεδρίες του Προεδρείου. Γεια σας και θα τα πούμε το απόγευμα.